Ε, ε, ε, συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρόλα αυτά έχουν ληφθεί περιοριστικά μέτρα για 28 άτομα που βρίσκονται στον κατάλογο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιράν. Ευχαριστώ τον Πίτρο Πονταλή. Έχουμε 7 ψηφίσματα και τώρα ε, εφόσον έληξε η συζήτηση θα υπάρξει η ε, ψηφοφορία. Καταρχήν ε, θα ψηφίσουμε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφαλείας στην περιοχή του Σαχέλ. Έχουμε 7 ψηφίσματα και ένα κοινό ψήφισμα από έξι πολιτικές ομάδες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην ψηφοφορία σχετικά με τις περιπτώσεις ατιμορρησίας στις Φιλιππίνες όπου πάλι έχουμε ένα ψήφισμα από πολλές πολιτικές ομάδες, 7 των αριθμών και ο συνάδελφος Σιλβέστρης ζήτησε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? τότε θα ψηφίσουμε ονομαστικά και τώρα εγώ ε, δεν έχω την ε, κάρτα μου αλλά είναι στη θέση μου. Ε, ξεκινά η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. στο 143-144 μπορείτε να ψηφίσετε για μένα παρακαλώ διότι βλέπετε ότι γίνεται κατόπιν δικιάς μου προτροπής. Ευχαριστώ. Ψηφίσατε όλοι. Α, χαίρομαι πολύ που μου φαίνεται την κάρτα μου. Ε, παρακαλώ ε, ε, να με συγχωρήσετε για αυτή την αναμπομπούλα και έτσι τώρα δεν κάνουμε τίποτα το παράνομο έχω και εγώ ψηφίσει ψηφίσατε όλοι λίγη ψηφοφορία ε, έχουμε 49 υπέρ και 3 κατά μετά εξετάζουμε την περίπτωση των, εθνοτι... των εθνοτικών μειοτήτων στο Ιράν όπου υπάρχουν επίσης ε, ε, ψηφίσματα πολλών πολιτικών ομάδων έχει αποσυρθεί η πρώτη τροπολογία και ξέρω ότι ο κύριος Πόσελ θέλει να κάνει μια προφορική τροπολογία. Εδώ μιλάμε για την διάρκεια. Ε, ε, για την διάκριση κατά των μη των μουσουλμάνων. Θα ήθελα εδώ να διευρυνθεί στους χριστιανούς και στις υπόλοιπες μειονότητες, γι' αυτό και προτείνουμε την ε, το διωγμό των πέραν των ασύρων και άλλων θρησκευτικών ομάδων δηλαδή να υπάρχουν και οι ασύροι αλλά και οι χριστιανοί ευχαριστώ έχει κάποιος αντίρρηση δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση κατόπιν αυτού Ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. και αυτή, αυτό το ψήφισμα έγινε σχεδόν ομόφωνα αποδεκτό με δύο μόνο αποχές. Η κυρία Ντεκάιζερ, ε, ε, εγώ εγώ ψήφισα και τράβηξα ίσως πολύ γρήγορα την κάρτα μου. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχει καταγραφεί η ψήφος μας. Θα το ελέγξουμε και θα δούμε στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, από το ε, ΕΛΚ και από το, τους σοσιαλιστές έχω λάβει τις εξής παρακλήσεις να τοποθετηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο κύριος Σούλμας, μεταφορών Άνταμ Κόσα και ε, Γεωργία σε Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, επιβεβαιώνονται αυτέ οι αλλαγέ. Το πρακτικά θα υιοθετηθούν στην επόμενη συνεδρίαση και